Po pierwsze zabierze głos pan poseł Peter Jar. Ο κύριο Πέτερ Γιάρ, πρώτο που θα λάβει τον λόγο από πλευρά του ΕΛΚ, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο να πω ότι για το χρονοδιάγραμμα περίοδων συνόδου 2017 θα ήθελα να είμαστε πιο θαραλέοι, λίγο περισσότερο θάρρος να είχαμε, ώστε συνεδριάσεις ε, στις ε, Βρυξέλλες ε, έναντι των συνεδριάσεων των Ολομελιών του Στρασβούργου να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση. Ελπίζω να έχουμε ευκαιρία με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου να συζητήσουμε τα προβλήματα εκτενώς. Λυπούμε ε, πραγματικά για το ότι δεν επετεύχθη αυτό. Ίσως μπορούμε να πετύχουμε κάποιες βελτιώσεις περαιτέρω στο μέλλον. Παράκλησή μου, όταν είμαστε εδώ σε Ολομέλειες στο Στρασβούργο να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας και να έχουμε και μία μείνει ολομέλεια για παράδειγμα στις Βρυξέλλες που θα μπορούσαμε να την αφήσουμε να διαγραφεί για να γίνει μια πλήρης ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ λέει και ο Σάνοτ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο μας, το Ηνωμένο Βασίλειο, επί 142 μέρες συνεδρίασε πέρσι και το επέκριναν δρυμύτατα που συνεδρίασε μόνο τόσες μέρες. Όμως εμείς στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, στην Ολομέλεια και τη Μήνη Ολομέλεια, συνεδριάζουμε για μόνο πέντε μέρες το μήνα και σε τρεις από αυτές τις μέρες μόνο ένα κομμάτι της ημέρα συνεδριάζουμε. Καταλήγουμε με συζητήσεις στο Κοινοβούλιο όπου τα μικρόφωνα κόβονται από τους ομιλητές μετά από 60-90 δευτερόλεπτα ή δύο λεπτά. Και δεν έχουμε κανέναν τρόπο να επεκτείνουμε τις απόψεις μας και να απαντήσουμε και να κάνουμε κανονικό έλεγχο προτινόμενης νομοθεσίας. Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο λογικό να έχουμε επαρκή χρόνο που θα μας διατίθεται για σωστή συζήτηση, η λογική συζήτηση και εκείνοι που πιστεύουν στις δομές και τα θεσμικά όργανα ε, θα πρέπει αυτό να το καλωσορίσουν. Νομίζω ότι τελειώσαν τα 60 δευτερόλεπτά μου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Άρνοτ. Ο κύριος Βαντάλεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό που γίνεται. Για το 2017 πρέπει να ψηφίσουμε χωρίς τροπολογίες. Και τώρα δεν γίνεται υπάρχουν επεξηγήσεις ψήφου για μια ψηφοφορία η οποία βασικά δεν μπορούσε να γίνει. Μα είναι εντελώ αντιδημοκρατικό αυτό. Με ακούτε. Μιλούσα πρόεδρε. Καλό θα ήταν να με ακούτε, να ακούτε τα επιχειρήματά μου. Έλεγα εγώ ότι έχουμε επεξηγήσεις ψήφου για μια ψηφοφορία που δεν έγινε βασικά. Δεν είναι δημοκρατικό. Η διάσκεψη των Προέδρων θα πρέπει να το δει. Θα πρέπει να μπορούμε να ψηφίσουμε αν υπάρχουν τροπολογίες, αλλά δεν μπορούσαν να υπάρχουν τροπολογίες. Δεν στέκει. Είναι ανόητο. Οι πρόεδροι των ομάδων θα πρέπει να το κοιτάξουν στη διάσκεψη των πρόεδρων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας προσέχω όταν ομιλείτε και παρεμβαίνετε. Πρέπει όμως να ακούσω και τις φωνές, ε, τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό το σημείο αναγράφει στην ημερήσια διάταξη προτού καταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση όπως αναφέρθηκε σε σχέση με τις ψηφοφορίες τώρα. Τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου περαιτέρω επεξηγήσει στην έκθεση της κυρίας, ε, έκθεσης της κυρίας Γκέριγκερ Όντενμπεργκ, Ευρωπαϊκής Διαδικασίας δηλαδή για τις μικροδιαφορές και διαδικασίες έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά Πρόεδρε. Θα ήθελα να δηλώσω ακριβώς γιατί αυτή την ευρωπαϊκή διαδικασία την υποστήριξα ψηφίζοντας υπέρ. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα αυτό όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και προστασία επίσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικά μέτρα διασυνοριακά όσον αφορά τις ε, Είναι μια ανάγκη που υπάρχει όταν αγοράζει κάποιο το διαδίκτυο. Ένα κλασικό παράδειγμα η επιστροφή χρημάτων όταν κάποιο εμπόρευμα είτε δεν παραδόθηκε έγκαιρα ή δεν παραδίδεται ή έχει κάποιες ελλείψεις. Ε, και τώρα σε σχέση με το ε, δεν γνωρίζουν κάποιοι άνθρωποι τις σχετικές λεπτομέρειες θα πρέπει να γίνει ένα βήμα δικαστικό ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις διεργασίες και να μην επιβαρύνονται γραφειοκρατικά ή μετέλη. Χαίρομαι ότι από 2 ε, σε 5.000 ευρώ αυξήθηκε παρότι ε, σε σχέση με την αύξηση μπορεί να είχαμε κάποιες άλλες επιθυμίες. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν θα πρέπει τα εργασιακά δικαιώματα να αποτελούν αποκλειστικό σημείο αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Το υποστήριξα και εγώ το αίτημα αυτό ως πρώην υπουργό Δικαιοσύνης στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Γνωρίζω πόσο μεγάλο και έντονο είναι το πρόβλημα των διασυνοριακών διαφορών. Πολλές επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες φοβούνται να ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία. Διαρκούν αυτές οι διεργασίες περισσότερο και είναι πιο δαπανηρές. Είναι καλό λοιπόν το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να άρει αυτά τα εμπόδια και προσκόμματα ώστε να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης που θα ανακουφίζει τους πολίτες. Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει αυτές οι διεργασίες με βιντεοδιασκέψεις να ε, πρικίζονται και να εξοπλίζονται ώστε να είναι δυνατόν οι πολίτες να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των δαπανηρών ε, διοικητικών και δικαστικών ε, δαπανών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθηνότερες, πιο προσιτές διαδικασίες. Είναι σημαντικό για τους πολίτες αυτό, διότι η μη επικοινωνούσα δικαστική εξουσία ουσία είναι πρόσκομα. Σα ευχαριστούμε. Τώρα θα έχετε εσεί τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Două regulamente din unul din 2006, unul din 2007 care reglementează procedurile mai scurte speciale pentru cererile cu valoare mică și Ευχαριστώ για τις αιτήσει αυτές και για την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία πληρωμών θέλω να μιλήσω. Είναι κάτι για να βοηθηθούν επιχειρηματίες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιταχύνεται η δικαστική διαδικασία. Εμείς εργαζόμαστε, ζούμε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς θα ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο. Αλλά θα έπρεπε να αλλάξουν οι κανονισμοί με τους εξής στόχους. Πρέπει να φτάσει το ποσό στα 5.000 ευρώ. Οι ηλεκτρονικοί μέθοδοι κοινοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι δικαστές επίσης θα πρέπει να μπορούν ο, κάθε φορά που γίνεται να χρησιμοποιούν τηλεδιασκέψεις και οι αποδείξεις θα πρέπει επίσης να δίνονται εξ αποστάσεως με τέτοιου είδους μέσα, τηλεδιασκέψεις δηλαδή και οι πληρωμές να γίνονται επίση εξ αποστάσεω. Όλα αυτά θα βοηθήσουν πολύ την εμπορική ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάρ. Ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μπορούσα να πω καλό είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Διεργασία για τις δικαστικές διεκδικήσεις διασυνοριακών θεμάτων που ήδη λειτουργεί η πείρα που είχαμε που ήταν θετική δείχνει ότι το κόστος ε, για τους εμπλεκόμενους μειώνεται κατά 40% και μειώνεται και η διάρκεια, η χρονική διάρκεια διευθέτησης των διαφορών. Και όλα αυτά σε σχέση με το 2.000 ευρώ, με την προσπάθεια να αυξηθεί σε 10.000 ευρώ, το ωραίο είναι με 10.000 ευρώ κατά 50% του συνόλου των διαφορών θα μπορούν ε, να διευθετούνται. Ιδιαίτερα προς όφελος των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν νομικές υπηρεσίες που μπορούν να διευθετούν τα θέματα των διεκδικήσεων. Όμως στην εσωτερική αγορά πρόκειται κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αν θα μπορούσαμε να έχουμε και περαιτέρω βελτιώσεις, αυτό θα ήταν πραγματικά κάτι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Danke sehr. deputats ε, Ο Μάμικινς. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται επί της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών, κρατών μελών και πολιτών. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία. Για, να, για την επίλυση των μικροδιαφορών, οι πολίτες πρέπει να δίνονται να προσφύγουν στο δικαστήριο. Κυρίως αν το θέμα αφορά οικονομική αποζημίωση. Πρέπει να υπάρχει εύρυθμο, αποτελεσματικό σύστημα για να διευθετεί τις μικροοικονομικές διαφορές. Η έκθεση εστιάζεται ακριβώς στην αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος για τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Και εγώ υπερψήφισα διότι υποστηρίζω πλήρως την πρόταση. Πιστεύω ότι μια αποτελεσματική διαδικασία επιλύσεως των μικροδιαφορών θα συμβάλλει στο να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο οικονομικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Πόλτσακ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω το πώς ψήφισα και γιατί την έκθεση αυτή την υποστήριξα και θεωρώ προσωπικά ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτού του δικαίου ενός σύνθετου πλαισίου διατάξεων που διασφαλίζουν το δικαίωμα των ατόμων να προσφύγουν σε δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη δικαστικά. Πρέπει όμως να είναι απλές αυτές οι διεργασίες και αυτή η πρόταση αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Η αξία, οριακή αξία 5.000 ευρώ είναι ένα μέγιστο κατόφλι ή ανόφλι θεωρώ και οι πολίτες ε, πρέπει να γνωρίζουν το τι συμβαίνει αυτό, αυτή η δυνατότητα ισχύει και υπάρχουν δυνατότητες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ε, δικαστικά. Οι ε, τα θέματα του κόστους είναι να αποτελούν βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε όμως να επικοινωνήσουμε καλύτερα, να γίνουν καλύτερα γνωστά στους πολίτες, ώστε να υπάρχει η πρόληψη που απουσιάζει εδώ για την έκθεση τώρα του κυρίου Άντζε Γκζίμπ περιορισμός εκπομπών ορισμένων ρήπων στην ατμόσφαιρα πρώτος που θα παρέμβει θα είναι η κυρία Μόνικα Μακαβέ ένα λεπτό παρακαλώ uh, Ευχαριστώ πρόεδρε η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η κύρια αιτία διαφόρων ασθενειών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εγκαταστάσεις παλιές για ηλεκτρισμό, για επιχειρήσεις και για κατοικίες και για θέρμανση, για τη βιομηχανία, με αποτέλεσμα διάφορες εκπομπές ρηπογόνων σωματιδίων. Κάπου 150.000 ε, όμως εγκαταστάσεις δεν ευθυγραμμίζονται προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με την σημερινή ψηφοφορία θα τηρηθούν τα όσα έχουν εγκριθεί και οι εγκαταστάσεις αυτές δεν θα ξεφεύγουν από την νομοθεσία και δεν θα ρηπαίνουν την ατμόσφαιρά μας, τον αέρα που αναπνέουμε, και που οδηγούν σε διάφορες ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου λοιπόν 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις ε, κατώτερες προδιαγραφές ε, ενέργειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αυτές για να δούμε τη συμμόρφωση προς τις κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίτερ Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οφείλω να πω ότι ψήφισα, υπερψήφισα την έκθεση, αλλά παρόλα αυτά δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι γιατί το μήνυμα είναι καλό μεν, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι τα όσα αναφέρει η έκθεση θα εφαρμοστούν. Για δύο λόγους υπερψήφισα. Πρώτον, γιατί λέει ότι με την ε, τροποποίηση που προτείνεται, η δυνατότητα εφαρμογή της οδηγίας βελτιώνεται. Άρα, θα έχουμε δηλαδή ένα πραγματικό εργαλείο για να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση της ατμόσφαιρας ε, χωρίς να επιβάλλουμε νέα βάρη στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν είναι ένα βήμα ε, να αποφύγουμε την γραφειοκρατία. Καλό λοιπόν αυτό. Και ζητάω από τους συναδέρφους της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να φροντίσουν ώστε όσα αναφέρονται στην έκθεση να τεθούν πράγματι σε εφαρμογή. Ευχαριστούμε. Μάμη κίνηση τώρα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Έχουμε την καθημερινή ζωή όπου χρησιμοποιούμε καθημερινά θέρμανση και ηλεκτρισμό. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Ούτε τα οικονομικά μας μοντέλα θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά. Ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι παράλληλα με αυτά έχουμε και τη ρήπανση της ατμόσφαιρας, δημιουργία σκόνης κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μόνο δύο οδηγίες. Την οδηγία την οικολογική, το eco-design και την οδηγία που αφορά τις μεγάλες εγκαταστάσεις ε, καύσης για να κάνουμε διαχωρισμό της παραγωγής ενέργειας από ρηκτά κάψιμα από τις μονάδες παραγωγής και μεταξύ των δύο οδηγιών και να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη όσον αφορά τα μέτρα θα ήθελα μια τρίτη οδηγία ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να αυξήσουμε όμως και σημαντικά το διοικητικό άχθος μέσω των μέτρων που θα θεσπίσουμε. Η κυρία Τζιλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση GRIPS διότι είναι πολύ σημαντική για το πακέτο και τον καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης να μειώσουμε τις εκπομπές που είναι επιβλαβείς και να πιώσουμε την ατμόσφαιρα και στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη έρευνα. Έρευνα πρόσφατη δείχνει ότι ο θάνατος λόγω μόλις της ατμοσφαίρας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο υψηλός από το 30.000 θανάτους που υπολογιζόταν σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη 500.000 άτομα πέθαναν πρώιμα σαν αποτέλεσμα της ρήπανσης του, της ατμόσφαιρας κάθε μέρα. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλο βάση της κοινωνίας και σε αυτό το πλαίσιο επίσης θέλω να πω δύο λόγια για τις εκπομπές, το σκάνδαλο της Volkswagen, τις εκπομπές του Diesel. Είναι εξωφρενικό λόγω της επιβλαβούς ε, συνέπειας για την υγεία των ανθρώπων. Για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που πληρώνουμε τη ζωή τους οι πολίτες για ποινική συμπεριφορά μεγάλων ομήλων που επιδιώκουν κέρδη παντιοτρόπος. πάση θυσία θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγχει αυτά τα θέματα. Η Volkswagen κατέστησε σαφές ότι το παρόν σύστημα στο οποίο η αυτοκινητομηχανία ε, αντιμετωπίζει τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς και επιλέγει που γίνονται οι δοκιμές είναι κάτι που δεν λειτουργεί. Uh, Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Έγκερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την έκθεση αυτή και θα καταψηφίσω κάθε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα, για την η απασχόληση. Εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης χάνονται σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε θα σταματήσετε. Πότε θα σταματήσετε με αυτήν την νομοθεσία η οποία κοστίζει σε απασχόληση. Και τι θα κάνουν οι άνθρωποι όταν χάνουν τη δουλειά τους σε τέτοιες κλάδους που χρειάζονται ειδικά προσόντα. Θα έπρεπε να εξηγήσουμε στον κόσμο που χάνει τη δουλειά του γιατί βρίσκεται σε αυτή την ε, κατάσταση και γιατί το κάνουμε. Για κοιτάξτε καλύτερα την κατάσταση που δημιουργείται, τη μιζέρια σε διάφορες κοινότητες τοπικές οι οποίες είχαν δουλειά και τώρα θα τη χάσουν έχετε δημιουργήσει μαζική απασχόληση προωθώντας τέτοια νομοθεσία που σκοτώνει και τις θέσεις απασχόλησης και την Βρετανική βιομηχανία. Ευχαριστούμε. Τώρα συνεχίζουμε και θέλω να ζητήσω από τους ομιλητές να λένε από πριν αν θέλουν να πάρουν το λόγο ω επεξήγηση ψήφου, γιατί έτσι οργανώνουμε καλύτερα τη δουλειά μα. Τέλο πάντων, ο κύριο Πόλτσακ το ζήτησε το λόγο, αλλά σα παρακαλώ να μα ενημερώνετε νωρίτερα αν θα παίρνετε το λόγο στην επεξήγηση ψήφου για να προετοιμάζουμε καλύτερα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την ανταπόκριση. Ζήτησα τον λόγο για το πρώτο σημείο. Δεν γνωρίζω γιατί δεν αναφαινόταν το όνομά μου σχετικά, αλλά πολύ σύντομα. Υποστήριξα την πρόταση. Όμως, σε σχέση με τη στάση μου ήμουν, κάποιο, ήμουν κάπως προβληματισμένος. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να δημιουργήσει ένα θετικό πλαίσιο δράσεων ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόβλημα των εκπομπών ρήπων Volks, οχημάτων Volkswagen βλέπουμε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Τα επόμενα προγράμματα θα πρέπει να μπορέσουν να λειτουργήσουν όταν θα γνωρίζουμε επακριβώς πώς οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές τηρούνται και με ποιο τρόπο εφαρμόζονται. Και πάλι ευχαριστώ Πρόεδρε για το ότι ανταποκριθήκατε στο αίτημά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Περνάμε στη συνέχεια στις επεξηγήσεις ψήφου όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Τζοβάνι Λαβία για τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Πρώτος που θα παρέμβει ο κύριος Άντρες Μανίκινς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι καζεΐνες, η καζεΐνη ανήκει σε μία ομάδα ουσιών που σχετίζεται με τις πρωτεΐνες που περιέχεται στο γάλα, τον ζωικό γάλα. Είναι φυσική ουσία, χημική, που βρίσκεται και στο ανθρώπινο σώμα, η καζεΐνη. Περιέχει αμινοεξέα που είναι σημαντικά για την πρωτεϊνική μας δίαιτα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις ουσίες. Πρέπει η νομοθεσία μας να προσαρμοστεί δεόντως για να ελέγχεται η διαθεσιμότητα των καζεϊνών και των καζεϊνικών αλάτων στη διεθνή αγορά. Κάτι άλλο που αφορά την τυποποίηση θα βοηθούσε τους καταναλωτές να καταλαβαίνουν πραγματικά τι τρόφιμα αγοράζουν. Και γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λέει κύριος Ποσπίσιλ πρόεδρε. Υποστήριξα το αίτημα. Με μια πρώτη ματιά μπορεί κανείς να πιστεύει ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη ρύθμιση που θα δυσκολέψει τη ζωή μας. Το αντίθετο όμως ισχύει πράγματι. Πιστεύω ότι η ενιοποίηση των προδιαγραφών θα αποτελέσει σαφή προσδιορισμό των ποσοστών υγρασίας και των άλλων συνιστοσών και θα οδηγηθούμε στο να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα γίνει προϋπόθεση και για, την, για τους διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις. Και αυτό θα είναι θετικό για τη βιομηχανία και τα εργοστάσια, για τους ε, ατομικούς, για τους επιμέρους καταναλωτές, διότι θα βελτιωθεί η ποιότητα, θα αναβαθμιστούν οι διαδικασίες ποιότητας και οι διατάξεις σχετικά με την ποιότητα και ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή θα άρουμε επίσης τα προσκόμματα στην ενιαία εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και η τελευταία επεξήγηση ψήφου σχετικά και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 3 η ώρα. Ευχαριστώ όλους σας.